Euh, Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς, με τις καταιγίδε υπάρχουν ε, πολύ λίγοι παριστάμενοι και υπάρχουν και πολλοί που θα φτάσουν με καθυστέρηση λόγω και ακυρώσεων πτήσεων. Οπότε ζητώ εξ ονόματός του συγγνώμη, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν πολλοί. Δεν είναι πολλοί που έχουν ήδη φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον κύριο Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, που είναι πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα ε, θα περάσω κάποια διδικαστικά το ένα έγκριση μερσία διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει. φαντάζομαι ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερσία διάταξη. Σημείο 2. ανακοινώσει. δεν έχω κάποια ανακοίνωση, οπότε προχωρώ αμέσω σημείο 3 την ανταλλαγή απόψεων, τον κύριο Σισιλιάνο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα πραγματικό πυλώνα ε, του Διεθνού Συστήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε γείτονες στο Στρασβούργο. Η υποεπιτροπή μας παρόλα αυτά σπάνια έχει το προνόμιο να έχει μια ανταλλαγή απόψεων με το δικαστήριο, παρότι η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία σίγουρα είναι κοινό ενδιαφέρον ε, και συμφωνούμε με την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, κάτι το οποίο συμμερίζονται τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης που γιορτάζει την 70η επέτειο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ε, πάνω από 20.000 αποφάσεις του δικαστηρίου που βελτίωσαν τη ζωή των ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο στην Ήπειρό μας και επίσης έχουν παράσχει και μία ακόμη ε, έμπνευση ώστε να ε, ψωθούν σε ανώτερο επίπεδο τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ε, σύμβαση μπορεί να μην είναι ένα νέο νομικό μέσο, αλλά έχει να λάβει και νέες προκλήσεις, παραδείγματος χάρη προστασία ιδιωτικής ζωής, δεδομένων ή βιοιατρική νέοι τομεί, αναδυόμενοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε το σύστημα τη σύμβαση με μεταρρυθμίσει, αλλά υπάρχουν προκλήσει, παραδείγματο χάρη η καθυστέρηση για την εκδίκαση υποθέσεων, η ανάγκη τη πλούσια εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου. Κάτι σημαντικό επιση ε, είναι η πρόσβαση τη ευρωπαικη ενωση στη Σύμβαση. Σίγουρα πολλά έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα, πολύ σημαντικό για εμά. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, να ακούσουμε για τις νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τον χώρο δικαιοσύνη και την άμεση γειτονία τη Ένωση, τι γίνεται μέσα παραδείγματο χάρη στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Τουρκία προφανώ και στην ε, Ανατολική γειτονία. Χαίρομαι ιδιαίτερω λοιπόν που μα δίνετε σήμερα η δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει μαζί σα ε, για τι διάφορε προκλήσει και το θετικό εκτιμένο του δικαστηρίου. Θα θέλαμε να ακούσουμε όμως και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σήμερα και πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερες γέφυρες μεταξύ Κοινοβουλίου και Δικαστήριου. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Κάνατε μία τέλεια εισαγωγή Πράγματι, κατάλαβα σωστά ότι θέλετε να ε, σας κάνω ένα γενικό απολογισμό της κατάστασης, να έχετε λίγο μια ιδέα του που βρισκόμαστε και εν συνεχεία είμαι στη διάθεσή σας ε, να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας και να εμβαθύνουμε στα διάφορα ζητήματα που και εσείς αναφέρατε. Πράγματι, η φετινή χρονιά είναι η 50η επέτειος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για τις επιτυχίες ε, του συστήματος αλλά και τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες του συστήματος. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ε, αποδείχθηκε ότι είναι ένα μοναδικό εργαλείο υπό την έννοια ότι ουσιαστικά έχει διεισδύσει σε όλους τους τομεί του διεθνούς δικαίου. Καμία κλασική άλλη Ευρωπαϊκή Σύμβαση δεν έχει καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα με την πολύ πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της τότε Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αφορά το ε, αστικό δίκαιο, τις δικονομικές διαδικασίες, ποινικό δίκαιο, ποινικές διαδικασίες, εμπορικό δίκαιο, εμπορικά σήματα, νέες τεχνολογίες, φυσικά δημόσιο ε, δίκαιο συνταγματικό, διοικητικό, ε, συντομία, είναι παρόν σε όλα τα μέτωπα. Και βέβαια αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε και είναι μεγάλη πρόκληση για τους νέους δικαστές του δικαστηρίου που όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα υποθέσεων που τότε όλων των κλάδων του διεθνούς δικαίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν πολλές υποθέσεις ε, που έχουν να κάνουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικώ το διεθνές δίκαιο και βέβαια και το συγκριτικό δίκαιο. Γιατί αν θέλουμε να αποφανθούμε επί αυτών θεμάτων, ενίοτε χρειάζεται να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη του δικαίου για να δούμε πού βρισκόμαστε πριν αποφανθούμε για τα διάφορα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Ο δεύτερο, δεύτερη πρόκληση επιτυχία, αν θέλετε, είναι το πώς θα είναι ένα ζωντανό εργαλείο αυτή η σύμβαση που μετά από 70 χρόνια ύπαρξης θα παραμείνει μοντέρνα. Και αυτό δεν είναι βέβαια εύκολο. Είναι ένα δόγμα, θέλετε, που έχουμε εισαγάγει αυτό του ζωντανού εργαλείου, ζωντανού νομικού μέσου από τη δεκαετία του 70 με την Βρετανική υπόθεση ε, κατά Ενωμένου Βασιλείου. Έκτοτε λέμε ότι αυτό το εργαλείο θα πρέπει να εννοείται ε, με βάση ε, τις καθημερινές σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης. Όχι απλά να δούμε ποια ήταν η βούληση των ιδρυτών πατέρων. Πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς αυτή η σύμβαση ε, συνεχή βάση για να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα και στις συνθήκες της σημερινές. Αυτή η ερμηνεία ε, φαινόταν επαναστατική τότε, τώρα δεν είναι. Είναι μια μέθοδος ερμηνεία στην οποία επικύρωσε και το ανώτατο, το Συνταγματικό Δικαστήριο των ε, κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και το Διεθνές Δικαστήριο, που είπε κάτι πολύ απλό, δηλαδή όταν έχουμε ένα νομικό μέσο που δεν έχει κάποιο περιορισμό προ τη διάρκεια του, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και όταν αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει όρου γενικού, ε, υποτίθεται ότι τα κράτη που είναι συμβαλόμενα έχουν τη βούληση να το ερνεύουν και να το εφαρμόζουν εξελικτικά, ώστε να παραμείνει επίκαιρο ε, όσο ε, παραμένει σε ισχύ. Τρίτη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι και επιτυχία ταυτόχρονα κατά την απόψη μου τουλάχιστον, είναι η εναρμόνιση, η πρόκληση της εναρμόνισης των ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε 47 κράτη-μέλη, 27 εξ αυτών είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πρότυπο πρέπει να ισχύει, ένα ενιαίο πρότυπο και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι πάντοτε εύκολο ή προφανές κάτι τέτοιο. Και βεβαίως ε, πρόκειται και για μία εφεύρεση δηλαδή τα περιθώρια εκτιμήσεων των κρατών μελών. Τα περιθώρια εκτιμήσεων των κρατών μελών είναι μια έννοια που δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των διαφόρων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωση, όχι με συγχωρείτε, του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλω να πω, που είναι συμβαλλόμενο μέρο στη σύμβαση. Βέβαια υπάρχουν και κάποια όρια σε αυτά τα περιθώρια. Και αυτά εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης τις οποίες επιλαμβάνεται το δικαστήριο στα οικονομικά ζητήματα. Λέμε ότι είναι ευρύ αυτά τα, ευραία αυτά τα περιθώρια. Όταν όμως μιλάμε παραδείγματος διακρίσεις σε λόγο φύλου, εκεί είναι πολύ περιορισμένα τα όρια και ε, τα περιθώρια και ε, χρειάζονται πολύ βάσιμοι λόγοι για να αιτιολογείται μια διαφοροποίηση λόγω φύλου ή σεξουαλικού ε, προσανατολισμού. Αυτή λοιπόν η έννοια περιθώρια εκτιμήσεων μας επιτρέπει χωρίς όμως να προδίδουμε και τις αρχές της σύμβασης, ε, να προσπαθούμε να ε, εναρμονίζουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα πρότυπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις ε, του θεσμού μας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων, πρώτα απ' όλα το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, Έχουμε ένα πρόβλημα με την καθυστέρηση τις εκδίκασης υποθέσεων έλαβα το 2011 είχαμε 60.000 ε, εκκρεμούσες υποθέσεις και με διάφορες μεταρρυθμίσεις, μάλλον ε, ήταν 160 και έχουμε ε, καταφέρει να μείνουμε στις 60.000 απορροφήσαμε, δηλαδή 100.000 και έχουμε επιληφθεί και νέων υποθέσεων. 40 με 45.000 υποθέσεις νέες το χρόνο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, στις διάφορες σχηματισμούς ε, με το μονοπρόσωπο τριμελές και ευρεία σύνθεσης ε, σώμα. Έχουμε λοιπόν αυτή την καθυστέρηση, αυτό το backlog που το απαρτίζουν συνήθως 20.000, κυρίως 20.000 υποθέσεις που δεν είναι επαναληπτικές, είναι ευρεία συνθέσεως που αφορούν ε, το βασικό πυρώνα, πυρήνα ε, και είναι σημαντικές υποθέσεις, άλλες είναι επαναλαμβανόμενες, επαναληπτικά θέματα. Και πολλές φορές μπορούν να λυθούν με είτε διμερή διακανονισμό, είτε με φιλικό διακανονισμό. Αλλά έχουμε αυτές τις 20.000 υποθέσεις που είναι ο σκληρός πυρήνας αυτού αυτή τη καθυστέρηση που άπτονται σημαντικών υποθέσεων και γι' αυτό και καθυστερούμε. Έχουν και μια άλλη πρόκληση ε, αυτή της εκτέλεσης. Ε, κατά γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε πω το ποσοστό εκτέλεσης ε, του δικαστήριου είναι ακρό ικανοποιητικό. Έχουμε τη βοήθεια από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. που είναι το μόνο διεθνέ όργανο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αυτό το σύστημα ούτε σε επίπεδο περιφερειακό, ούτε σε επίπεδο οικουμενικό υπάρχει ένα ανάλογο σύστημα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πλέον στη ότι αυτή η Επιτροπή, ε, Επιτροπή Υπουργών είναι ένα διπλωματικό πολιτικό όργανο που δεν υπάρχει πιθανά αλλού. Άρα το σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μοναδικό και σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο η Επιτροπή Υπουργών, που έχει την βασική ευθύνη και αρμοδιότητα για την ε, παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων. Υπάρχει και κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και ε, Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που εργάζονται σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης και σε εθνικό επίπεδο τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία έχουν συγκροτήσει εθνικές ατοικοκεπιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Βουλή των Ελλήνων. Την προσεχή τρίτη συγκεκριμένα ε, θα απευθυνθώ στην τροπή αρμόδια του ε, σε Βουλή των Ελλήνων που θα ε, θέσει ερωτήματα για την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν την Ελλάδα. Και τηρούμε των αλογιών αντίστοιχε επιτροπέ υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλα τα κοινοβούλια σχεδόν. Είναι κάτι πολύτιμο για εμά. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί βέβαια. Θα μπορούσα να αναφέρω όπως είναι η εθνικοί για την προσέγγιση των η συνήγορη του πολίτη κτλ. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας δώσω να καταλάβετε την πολυπλοκότητα του συστήματος ε, ε, είτε σε επίπεδο Συμβουλίου Ευρώπης είτε σε επίπεδο κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μία άλλη επιτυχία και πρόκληση είναι ο διάλογος. Διάλογος καταρχήν με τα ανώτατα και ανώτερα δικαστήρια. Γιατί ειδικά με αυτά. Επειδή πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να προσφύγει σε εγχώρια ένδικα μέσα και γι' αυτό οι προσφυγές που φτάνουν σε εμάς εξετάστηκαν από ένα ανώτατο συνήθως συνταγματικό δικαστήριο στο κράτος μέλος. Αυτοί είναι οι βασικοί μας συνομιλητές. Γι' αυτό εδώ και πέντε χρόνια έχουμε ένα δίκτυο ανωτάτων ε, ε, δικαστηρίων όπου συμμετέχουν 88 δικαστηρία των 38 χωρών μελών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο και θα θέλαμε να είναι αποτελεσματικό όχι μόνο ως προς την ανταλλαγή ε, πληροφοριών αλλά και σε μία συνομιλία δύο φορές ε, το χρόνο. Η ε, Γαλλική Προεδρία στις 12-13 Σεπτεμβρίου πέρσι διοργάνωσε μία συνάντηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος Μακρόν μας ε, υποδέχτηκε στα Ελίσια Παιδεία και προώθησε αυτή τη μορφή διαλόγου. Ο διάλογος δεν γίνεται μόνο με τα ανώτατα δικαστήρια, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Μπορώ να πω ότι ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, είναι επιτυχής, ε, γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή και περισσότερες φορές. Στις 21 Οκτωβρίου έγινε η τελευταία συνάντηση και πάντα επιλέγουμε το θέμα όπου εστιάζουμε την προσοχή μας. Υπάρχει ένας δικαστής από τη δική μας πλευρά και ένας από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στη συνέχεια προωθείται διάλογος μεταξύ δικαιοδοσιών. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι άκρος ενδιαφέρουσα και αποδοτική. Την ε, Τελευταία φορά ήρθαν εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου εδώ και νομίζω ότι ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι από αυτή την συνεργασία. Βεβαίως μας ενδιαφέρει και το θέμα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, με το 14ο πρωτόκολλο δώσαμε πράσινο φως, εγκρίθηκε το 2004 και τότε Απλώς αναφερόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από πλευράς λοιπόν Συμβουλίου της Ευρώπης με το 14ο πρωτόκολλο έχουμε εκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας επίσης προώθησε αυτή την προσχώρηση μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά και στη συνέχεια μάλλον στις 24 Μαρτίου θα ξαναρχίσουμε αυτές τις συζητήσεις μετά από την επιστολή που προσυπέγραψαν ε, οι κύριοι Γιούνκερ Τίμπερμανς και η Γενική Γραμματέας του ΕΔΑΔ, η κυρία Μπούτσιτς. Στις 18 ε, 8 Νοεμβρίου με τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθήσαμε να δούμε πώς έχει κατάσταση, πώς έχει εξελιχθεί. Είμαι αισιόδοξο γιατί ξέρω ότι υπάρχει μία νέα όθηση επί του θέματος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί βεβαίως, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούρου και δεν θα πρέπει να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιφυλάξεις από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διαδικασία της κύρωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα επιδέξιοι, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο για να λάβουμε υπόψη και τις επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να μην δημιουργήσει άνηση μεταχείριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, θα φτάσω στο τελευταίο θέμα παρουσίαση σε σχέση με τις προκλήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Βλέπω τέσσερις προκλήσεις την πρώτη την αναφέρατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε. Είναι η μετανάστευση, το θέμα της μετανάστευσης. Και αυτό ως προς τους ετούντες άσυλο. Έχουμε πολλές προσφυγές κατά της Ελλάδας, όπως φαντάζεστε, κατά της Ιταλίας επίσης και έχουμε και μία υπόθεση κατά του Βελγίου που αυτή τη στιγμή εκρεμεί ενώπιον της ε, Ολομελίας μας κατά της Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και των σκανδιναβικών χωρών. Πρόκειται λοιπόν για αρκετές χώρες συμβαλόμενα μέλη Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την Νότια Ευρώπη, αλλά και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης και ε, πρόσφατα ελήφθη μια απόφαση κατά της ε, Ρωσίας και, Ρωσίας και κατά της ε, Ουγγαρίας ως προς το κλείσιμο της οδού των Βαλκανίων και φυσικά και τις συλλογικές ε, εκδόσεις όπου αποφανθήκαμε κατά της Ισπανίας. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση σε σχέση βεβαίως και με τους ενάγοντες πρωτίστως. Ποιες είναι τώρα, ποιοι είναι οι βασικοί μας άξονες για να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε την κατάσταση. Τρεις είναι οι άξονες. Καταρχήν, να κρατήσουμε το δικαιοδοτικό και εκτιμένο τη σύμβαση της Γενέβης για, για το καθεστώς των προσφύγων. Επίσης, το ρυθμιστικό και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας την ανάγκη να ξαναδούμε την Συμφωνία του Δουβλίνου και ο τρίτος άξονας της νομολογίας μας είναι να θέσουμε τα ε, στάδια της ε, διαδικασίας που αφορά τις μεταναστευτικές ροές για να μην γίνονται ε, συλλογικές εκδόσεις. Το δεύτερο βασικό ζήτημα σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη είναι το δημοκρατικό έλλειμμα. Υπάρχουν υποθέσεις που φτάνουν ως εμάς και αφορούν το θέμα της αμεροληψίας των δικαστηρίων. Έχουμε υποθέσεις κατά της Ρουμανίας, της ε, Πολωνίας. Έχουμε και μια μεγάλη υπόθεση κατά της Ουγγαρίας και εδώ βάζουμε άλλον έναν κρίκο στη νομοθεσία μας και υπήρξε και μία υπόθεση, παρόμοια υπόθεση στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, υπόθεση κατά της Πολωνίας. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 18 της Σύμβασης, ε, μιλάμε για παρέλκυση ε, εξουσιών. Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 18 και 19. Ενεργοποιήθηκε αρκετές φορές κατά της Τουρκίας, Αζερβαϊτζάν, Ομοσπονδίας της Ρωσίας κλπ. Για να ε, καταδείξουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το κράτος δικαίου όπου πραγματικά υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Ένα άλλο θέμα που επανέρχεται αφορά την τρομοκρατία, τις υποθέσεις κατά της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ε, υποδίκους, είτε θύματα τρομοκρατίας ή τρίτες χώρες, μάλλον ε, κάτοικοι τριών τρίτων χωρών που θεωρούνται ε, θύματα τρομοκρατίας. Έχουμε το Big Brother Watch κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, πρόκειται για μέτρα τα οποία έλαβε η MI6, η μυστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, με βάση την υποκλοπή ενός τρεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων Πρόκειται για θέμα εθνικής ε, κυριαρχίας. Υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που αφορά τη Σουηδία με παρόμοιο περιεχόμενο και εκρεμούν ενώπιον της ολομελίας μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο κανόνας ο οποίος θα δεσπόζει και θα επικρατεί ως προς τις μυστικές υπηρεσίες. Ε, τέλος, η τέταρτη πρόκληση αφορά ένα 15% των υποθέσεων μας και είναι ε, ε, διακρατικές υποθέσεις ή ε, μεμονωμένες υποθέσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του συστήματος έχουμε οκτώ τέτοιες διακρατικές υποθέσεις, Ουκρανία κατά Ρωσίας, η υπόθεση της Κρυμαίας, όπου έγινε ακροαματική διαδικασία. Έχουμε και την υπόθεση Ντόμπας και άλλες τρεις υποθέσεις, αλλά πάντα ε, διακρατικές, κυρίως Ουκρανία κατά Ρωσίας. Επίσης, Γεωργία κατά Ομοσπονδίας της Ρωσίας και μία υπόθεση όπου ελήφθη ήδη απόφαση είναι η δεύτερη τέτοιου είδους και μια τρίτη υπόθεση η οποία θα κριθεί τώρα. Και επίσης υπόθεση Σλοβανίας, Σλοβενίας κατά Κροατίας που έχει περισσότερο οικονομικό περιεχόμενο αφορά τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος καθώς και την, ε, τα δικαιώματα των εναγωμένων σε σχέση με το τραπεζικό δίκαιο. Ε, εδώ μπορώ να πω ότι υπάρχουν και πολλές μεμονωμένες ε, υποθέσεις ως προς τον Αγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Αυτές οι υποθέσεις μας απασχολούν ιδιαίτερα διότι πίσω από αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν ζητήματα πολιτικής υφής. Βεβαίως το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το, τη δική του εντολή, δηλαδή δεν θα υπερβεί αυτή την εντολή, κρίνει τα ζητήματα από καθαρά δικαστική πλευρά, γιατί πολλές φορές και το ανώτατο ποινικό δικαστήριο, όπως ξέρετε, γνωρίζει το ίδιο θέμα. Πρόκειται για υποθέσεις που άπτονται πολιτικών ζητημάτων, αλλά το δικαστήριο περιορίζεται στην δική του εντολή, την οποία δεν υπερβαίνει. Αυτά, ε, κυρία Πρόεδρε, εντάχει σε σχέση με τις προκλήσεις, τα ζητήματα που μας απασχολούν και τις επιτυχίες μας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στα παρόντα μέλη. Ιζαμπέλ Πισλέρ, παρακαλώ, πρώτη, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επεκταθήκατε σε έναν πολύ ευρύ τομέα ε, και ήταν πολύ βοηθητικά τα σχόλια και οι εξήγησή σας. Έχω δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Καταρχάς παίρνω το λόγο να σας ευχαριστήσω θερμά αυτό είναι ο βασικός λόγος. Μιλήσατε όμως και για τις προκλήσεις ε, στο θέμα της βιοηθικής. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο. Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά που είπατε για αυτό το θέμα και με ενδιαφέρουν και τα λεγόμενά σας για τη μετανάστευση. Η πρόκληση είναι τεράστια που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ευρώπη και αν όχι την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη νομίζω έχουμε αποστολή στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα μεταβούμε τόπου να δούμε τι κάνουν εκεί και τι γίνεται εκεί με την υποεπιτροπή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δούμε πώς ε, ε, λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη, για να μην τα βλέπουμε μόνο από μακριά και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Αυτά τα δύο θέματα θέλω να αναπτύξετε δηλαδή και επίσης να σας πω και το τρίτο που με ενδιαφέρει. Υπάρχει το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και υπάρχει και το δικό σας δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Στρασβούργο. Ίσως το εξηγήσατε και δεν το κατάλαβα καλά. Έχετε κοινέ υποθέσεις, μπορεί να συμβεί αυτό, μια, την ίδια υπόθεση να την εξετάσει το δικό σας δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία, τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ιζαμπέλ Σάντο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον προσκεκλημένα μας, να ζητήσω συγνώμη γιατί έφτασα με λίγη ε, καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσω την ομιλία μου στην Ολομέλεια. Άκουσα ένα μεγάλο μέρος ε, της εισαγωγής σας, της παρουσίασης και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο και της προκλήσεις του δικαστηρίου σας σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Βρέθηκα στην Κροατία και τη Βοσνία την προηγούμενη εβδομάδα και ασχολήθηκα με μία από τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αναφερθήκατε σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Πρόκειται για ένα τρομακτικό σενάριο ε, άκρα της βίας της κροατικής αστυνομίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών που ήθελαν να μεταβούν από την ε, Βοσνία στην Κροατία. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ε, διερευνάτε το γεγονός, γιατί είναι ένα γεγονός μεγάλης εμβέλειας. Ε, ε πολλές οργανώσεις, πολλές ΜΚΟ έχουν προβάλλει και στοιχεία για την άκρατη βία της κροατικής αστυνομίας κατά των προσφύγων. Το κροατικό κράτος δεν δέχεται να διενεργηθεί έρευνα δυνάμει του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυσικά και μπορώ να σας πω ότι η μεταχείριση είναι απάνθρωπη και στιγνή, απαράδεκτη από την κροατική αστυνομία. Δηλαδή τους αποσπούν όλα τους, ό,τι έχουν, ό,τι έχουν και δεν έχουν, όλα τους, ας το πούμε, όλα τους τα περιοσιακά στοιχεία, ακόμα και τα παπούτσια τους αφαιρούν και τους αναγκάζουν να διασχίσουν το δάσος σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Εγώ έχω εικόνες που μπορώ να σας, φωτογραφίες που μπορώ να σας διαβιβάσω για τις απάνθρωπες συνθήκες προέκυψαν και θάνατοι ακόμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο ε, προβλέπετε κάποια διαδικασία παρέμβασης επί του θέματος έτσι ώστε να εγγυηθεί θούμε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλες τις χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Ιάννα, παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω. Πρώτον, για την κατάσταση στην Τουρκία. Από το πήμα του 2016 στην Τουρκία έχει απορρίψει το δικαστήριο διάφορες υποθέσεις υπό θεωρώντας ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα και ε, θεωρείται ότι το τουρκικό συνταγματικό δικαστήριο αποτελεί αποτελεσματικό μέσο επιδιόρθωσης της κατάστασης και είναι προσβάσιμο και παραμένει προσβάσιμο. Όμως, μετά από τις εσωτερικές εξελίξεις και το πραξικόπημα, η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού δικαστικού συστήματος στην Τουρκία είναι υπό αμφισβήτηση και δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη ε, σε αυτό το δικαστικό σύστημα. Επομένως, ερωτώ, το δικαστήριο του Στρασβούργου θα αναθεωρήσει την άποψή του για το, αν, για το ποια θεωρεί αποτελεσματικά εσωτερικά ένδικα μέσα στη Τουρκία. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσει την άποψή του μετά το πραξικόπημα του 16 και θέλω και να αναφερθώ και στα ονόματα, τα δύο πολύ γνωστά ονόματα των δύο εγκλήσεων εδώ και χρόνια στις τουρκικές φυλακές και γνωρίζετε την υπόθεση. Αυτό καταρχάς. Ε, κατά δεύτερον, τελευταία χρόνια είδαμε όλο και περισσότερες ε, υποθέσεις να υποβάλλονται ε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ποιο βαθμό λοιπόν έχει ασχοληθεί το δικαστήριό σας με τέτοιου είδους υποθέσεις. Περιμένετε όλο και περισσότερες να είναι τέτοιας φύσης και πώς σκοπεύετε να τις ε, αντιμετωπίσετε και να τις χειριστείτε. Ευχαριστώ εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Το Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων για πρώτη φορά θα ασχοληθεί με τον επαναπατρισμό ε, σε ένα κράτος μέλος. Δύο παππούδες πήγαν στο δικαστήριο και θέλουν η Γαλλία να επιστρέψει την κόρη της την κόρη Δεν είναι συνηθισμένες αυτές οι περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ περίπλοκες σε ηθικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο. Όμως είναι στο επίκεντρο οι υποθέσεις αυτές του τι εστί εθνική αρμοδιότητα, τι σημαίνει το να είσαι υπήκο συγκεκριμένη χώρα, τι σημαίνει εθνική κυριαρχία. Ορισμένοι έχουν προβάλει το εξή επιχείρημα. Δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση να καθοδηγείται από βραχυπρόθεσμους κινδύνους ασφαλείας ή από βραχυπρόθεσμες επιδιώξει που θα ικανοποιήσουν το εκλογικό σώμα. Θα πρέπει να έχει ε, ε, να βλέπει προς το μέλλον. Έχουμε φόβους, πολύ λογικούς φόβους των Ευρωπαίων πολιτών. Οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη προς την κοινωνία και να ακούσουν τις νόμικες ανησυχίες των πολιτών όταν έχουμε να κάνουμε με ξένους πατέρες. Δεν θα πρέπει να επιστρέφει κάποιος ο οποίος θέλει να ε, γίνει τρομοκράτης και μαχητής, ε, ξένους μαχητές. Και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να ασχολούνται με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Ε, ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Ε, ευχαριστούμε. Η Διάννα παρακαλώ. Για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε κύριε Σισιλιάνε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Μιλήσατε για την εναρμόνιση των κρατών, για το γεγονός ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη ξεκινούν να αξιοποιούν το δικό τους μηχανισμό, έτσι ώστε να αποφύγουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χθες το Europa Press μίλησε, ανέφερε ένα πολύ ανησυχητικό νέο Έχουμε το συνταγματικό δικαστήριο το Ισπανικό και οι δικαστές εκεί υιοθέτησαν την εξή στρατηγική να μπλοκάρουν την πρόσβαση των καταλωνών πολιτικών ε, κρατουμένων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή δέχτηκαν όλες τις προσφυγές για να μπορούν στη συνέχεια να τις ε, καθυστερούν και να τις βάλουν σε ένα σιρτάρι έτσι ώστε να μην εξαντληθούν τα εσωτερικά ενδοϊκά μέσα και να μην μπορεί η υπεράσπιση τους να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτού εκδικαστεί οριστικά και τεσσελεσιδικής η υπόθεση των επικεφαλής. Και άρα ε, βλέπετε ότι οι αιτήσει ανέρεσης ε, κινούνται στο 1% γενικά. Στην περίπτωση ε, γίνονται δεκτές, ενώ στο οι αιτήσει να ασχοληθεί το ανώτατο Ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο για τα θέματα αυτά συνήθως γίνονται δεκτές κατά 1% αλλά για τους πολιτικούς κρατούμενους τους Καταλανούς γίνονται δεκτές το 100% και έχουν γίνει και απεργίες πίνες, και πάρα πολλές ε, διαμαρτυρίες. Το Νοέμβριο ο, έγινε προσφυγή του Οριόλ Γιουνκέρας μετά από δύο χρόνια αναμονής. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για τη στάση των Ισπανών δικαστών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει μηχανισμό για να ανοιχνεύσει και να επιδιορθώσει τέτοιου είδους πρακτικές εσωτερικών δικαστηρίων που κάνουν τα πάντα για να παρακολύσουν την προσφυγή των ατόμων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πώς μπορεί να γίνει ε, πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο για να μπορέσει να επιληφθεί το συντομότερο ε, σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριος Κυμπουρόπουλος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας και μας ε, ε, αναφέρατε όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ πηγαία, πιστεύω, για μια Ευρώπη την οποία θέλουμε να είναι Ευρώπη ίσων, Ευρώπη πολιτών, Ευρώπη της κοινωνίας. Και μερικές φορές δεν, το πείτε, δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Ε, εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς πιστεύετε εσείς από που είστε ε, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η εξομάλωση των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλα τα ε, κράτη-μέλη και όλοι, όλα τα κράτη-μέλη να αναγνωρίζουν με τον ίδιο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα σέβονται, να τα τηρούν και να πάμε σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά όπως έχει επιτευχθεί μια οικονομική ένωση να επιτευχθεί και μια ένωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Σας ευχαριστώ. Ναι, θα σα δώσω δυνατότητα απαντήστε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Αν μου επιτρέπετε, έχω και εγώ να προσθέσω κάποιε δικέ μου ερωτήσει. Η πρώτη αφορά ε, την, ε, τον αντίκτυπο της αποχώρησης των Βρετανών, ε, πώς έχετε προετοιμαστεί και τι θα συμβεί σε επίπεδο δικαστηρίου. Δεύτερη ερώτηση, ποιος είναι ο αντίκτυπος της πρόσβασης στη συνθήκη. Είπατε ότι οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών ε, που είναι συμβαλόμενα στην σύμβαση είναι κάτι σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, τι ρόλο πιστεύετε ότι έχει να διαδραματίσει και το τρίτο ερώτημα, ξέρω ότι είχατε κάποιες υποθέσεις ε, πάνω σε ένα πολύ σημαντικό και λεπτό θέμα, ευαίσθητο θέμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η πρόσβαση στην άμβλωση. Και έχουμε υποθέσει την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και ιδίως Πρόκειται για την αποζημίωση, καταβολή αποζημίωση σε γυναίκε που δεν είχαν πρόσβαση στην άβλωση λόγω των πολύ αυστηρών όρων και προποθέσεων τη εθνική νομοθεσία. Αυτό έχει δημιουργήσει νομολογία που επιτρέπει ενδεχομένως την επανεξέταση της θέσης αυτής που δεν είναι ιδεολογική και θρησκευτική αλλά μπορεί να ερμηνευθεί κυρίως ως ζήτημα που άπτεται στην αξιοπρέπεια και την υγεία των γυναικών και που συνιστά αυτή η μη πρόσβαση στην άβλωση ε, σε διακριτική μεταχείριση. Όταν μια γυναίκα δεν έχει την ελεύθερη πρόσβαση, ουσιαστικά ε, δέχεται πλήγμα και ίδια της η ζωή, όπως είχαμε μια περίπτωση στην Ιρλανδία και πραγματικά ε, θα ήθελα να μου πείτε εσείς αυτό το θέμα πώς το λαμβάνετε υπόψη σε επίπεδο δικαστήριο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Τα στήματα βιοηθικής. Πράγματι είναι πολλά. Είχαμε ερωτήσει ε, για το τέλος της ζωής, υπόθεση Λαμπέρ για παράδειγμα, κατά ε, Γαλλίας. ή για τη βιοιατρική, για τα βιοιατρικά πειράματα. Τη συγκατάθεση σε ιατρικές επεμβάσεις ε, και τα λοιπά. Είχαμε θέματα για τις παρένθετες μητέρες. Ε, είχαμε μια συμβουλευτική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος του Γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, μάλλον ακυρωτικού δικαστηρίου. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, δείχνει πόσο καλή είναι αυτή η προσέγγιση δυνάμει του πρωτοκόλου 16 ε, που επιτρέπει στα ανώτατα δικαστήρια να θέτουν ερωτήματα για συμβουλευτικούς σκοπούς και ακολούθησε τις συστάσεις το Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο πλαίσιο της στάσης του δικού μας δικαστηρίου και υπάρχει και το άρθρο 7 της Σύμβασης του Βιέδο ε, για τη βιοιατρική η διεθνή, δηλαδή κατεξοχήν διεθνή σύμβαση για τα θέματα τη ε, βιοθική, πολύ λεπτά θέματα, από τον οποίο θα πρέπει να αποφανθούμε. Η σύμβαση του Οβιέδο για τη βιοτρική και τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέπει ε, στην Επιτροπή Βιοηθικής και στα συμβαλόμενα 30 τον αριθμό κράτη-μέλη, των οποίων τα πιο πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέτουν ερωτήματα και να διατυπώνουν αιτήματα ε, συμβουλευτικού χαρακτήρα ε, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δεν είναι αρμόδιο μόνο για τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά κατά κάποιο τρόπο και για αυτή τη σύμβαση του Οβιέδο για τη βιοιατρική. Αυτό θα είναι και μία πρεμιέρα αν θέλετε, ένα ιστορικό βήμα θα το χαρακτήριζα. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφαίνεται μόνο επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, άρα θα είναι η πρώτη φορά που θα αποφανθεί επί τη βάση μιας άλλης σύμβασης, τη σύμβαση της βιοηθικής. Αυτή τη στιγμή, ήδη σήμερα, δεν ενημερώθηκα πριν έρθω εδώ, δεν είχα το χρόνο, αλλά ήδη σήμερα η Επιτροπή για τον κανονισμό θα έπρεπε να θετήσει νέους κανόνες ώστε να μπορούμε να επιληφθούμε αυτού του αιτήματο που μόλις λάβαμε και αυτό θα γίνει άμεσα, αμελητή και ελπίζω μέσα στη χρονιά αυτή να είναι αυτή η πρώτη ευκαιρία να δώσουμε συμβουλευτική γνώμη για ε, την βιοετρική με βάση τη σύμβαση του Βιέδο. Βεβαίως πρόκειται για πάρα πολύ πλούσιο τομέα που άπτεται κυρίως του άρθρου 8 της Σύμβασης, ιδιωτική ζωή, οικογενειακή ζωή, αλλά και του άρθρου 2 που είναι το δικαίωμα στη ζωή, τέλος, αρχή ζωής κτλ. Και αυτό έρχεται να ε, συσχετιστεί και με τα ζητήματα περιάμβλωσης, τα οποία θα επανέλθω. Για τη μετανάστευση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ταυτόχρονα στην κυρία Σάντος. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ε, τα ε, προληπτικά μέτρα με βάση το άρθρο 39 του κανονισμού. Ασφαλιστικά μέτρα θα τα χαρακτήριζα. Είναι μια άμεση αντίδραση ε, Είμαστε ανοιχτοί 360 μέρες το χρόνο. 20 ώρες το 24ωρο για το κοινό. Για να λάβουμε ε, τις αιτήσει ασφαλιστικών μέτρων έχουμε δύο δικαστές ε, οι οποίοι ε, φημερεύουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και μπορούν να κληθούν να απαντήσουν σε τέτοια αιτήματα κατεπηγόντως. Υπάρχει ένα σύστημα checklist από τη γραμματεία και μια ειδική μονάδα ε, που πραγματικά δουλεύει με το χρονόμετρο, με το ρολόι. Οι εθνικοί δικαστές πολλές φορές καλούνται να δώσουν και γνωμοδότηση ε, στους εφημερίδες δικαστές μέσα στις επόμενες ώρες από την υποβολή ενός αιτήματος. Προείδρευα ε, σε ένα τμήμα ευρεία σύνθεση και έλαβα στο κινητό μου ένα μήνυμα που λέει «Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μας πείτε μέσα στο επόμενο μισάρο την άποψη για το τάδε θέμα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, χρειάστηκε να διακόψω τι εργασίε ε, του σώματος για να απαντήσω, να γνωμοδοτήσω σε εθνικό δικαστή, γιατί είναι θέμα που αφορούσε τη δική μου χώρα, την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που είναι σε ένα διάδρομο του αεροδρομίου και του απελάβνουν, για να επανέλθω σε κάτι το οποίο είπατε, σε ένα διαφορετικό βέβαια πλαίσιο, αλλά είναι μια πολύ επίγουσα κατάσταση και προσπαθούμε με τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα, ε, τα προσωρινά μέτρα, προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, δεν λέω ότι μπορούμε να λύσουμε τα υπαρξιακά προβλήματα της Ευρώπης, αλλά κάθε μέρα Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στις επάλξεις, να αφουγκραζόμεστα και να δίνουμε απαντήσεις το συντομότερο δυνατό όταν έχουμε να κάνουμε με κατεπήγοντα ζητήματα που άπτονται του δικαίωμα της ζωής, ακαιρεότητας ε, του προσώπου, όταν μιλάμε για άτομα τα οποία κινδυνεύουν να απελαθούν σε κράτη εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε κράτη που έχουμε εμπόλεμες συγκρούσεις. Η συνάδελφό σας στο βάθος, κυρία Κάνκο, αν βλέπω καλά, αναφέρθηκε πριν. Είναι λοιπόν ένα μέσο στο, το οποίο έχουμε στη διάθεση μας. Για να σας δώσω έτσι και κάποια ποσοτικά στοιχεία. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις χρειάστηκε να απαντήσω ως εθνικός δικαστής, μάλλον όχι να ε, απαντήσω, να δώσω μια άποψη, μια γνώμη για το εφημένο δικαστή αυτός που θα απαντήσει. Απλά μου ζητήθηκε η γνώμη μου σε 11 αιτήματα για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 11 αιτήματα μέσα σε 5 μέρες που αφορούσαν μόνο την Ελλάδα για να καταλάβετε λίγο πολύ την τάξη μεγέθους και τη σημασία του εργαλείου αυτού που είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα έχουμε δεκάδες επί δεκάδων αποφάσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών, για υποθέσεις ε, μεταχείρισης ε, στη σύλληψη ε, και την προσπάθεια απομάκρυσης, για το αν είναι νόμιμη ή μη κράτηση με βάση το άρθρο 5 της Σύμβασης και βέβαια και επί των συλλογικών μαζικών απελάσεων. Θα έχουμε σύντομα, μεθαύριο συγκεκριμένα, μια απόφαση για την Ισπανία. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν, οι απελάσεις, οι συλλήψεις, συνθήκες κράτησης, νομιμότητα κράτησης, οι μαζικές απελάσεις είναι αντικείμενο των αποφάσεων που άπτονται σε αυτό το ζήτημα της μετανάστευσης. Και συν ασφαλιστικά μέτρα που ανέφερε. Πανέρχομαι στο δικό σας ερώτημα. Αν δηλαδή Μπορεί ένα ερώτημα ε, ή ένα ζήτημα να είναι αντικείμενο εξέτασης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων και στο ε, ΔΕΚ ε, είναι η λεγόμενη υπόθεση Μπόσφορου, ε, Βόσπορος, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο. Ουσιαστικά είναι η ίδια υπόθεση που αφορά τη σχέση μεταξύ του συστήματος των ΗΕ, Εθνών, του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος της Σύμβασης. Πρόκειται για κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίε μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κανονισμού της Ένωσης ε, και εν συνεχεία η ίδια υπόθεση ε, που έκριναν οι δικαστές του Λουξεμβούργου ήρθε σε εμάς ε, δυνάμει της Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωματών. Μιλάμε για την αλληλεπίδραση τριών συστημάτων του παγκόσμιου που είναι τα, αυτό του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού που είναι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και το δικό μας στο και προσπαθούμε να καταλήξουμε εδώ σε αρμονισμένη ε, προσέγγιση. Στην προκειμένη υπόθεση έχουμε το τεκμήριο ισοδυναμίας ή αντιστοιχίας ότι δηλαδή παρέχεται ε, ισοδύναμη ε, προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή που ε, κατοχυρώ τη Σύμβαση την Ευρωπαϊκή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό για να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τη δουλειά μας με τους συναδέλφους από το Λουξεμβούργο. Έρχομαι στις ερωτήσεις της κυρίας Νόιμαν για την Τουρκία συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζετε πως μετά το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος ε, του Ιουλίου 2016, λάβαμε μέσα σε ένα μήνα 32.000 ε, περίπου υποθέσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί ένα τέτοιο όγκο υποθέσεων. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πράγματι δεν θελήσαμε εκείνη τη στιγμή να πούμε ότι το τουρκικό συνταγματικό δικαστήριο δεν είναι ε, ένα αποτελεσματικό ενδικό μέσο προσφύγης σε αυτό το δικαστήριο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ε, γνωρίζουμε, να γνωρίζετε ότι επιλαμβανόμεθα αυτών των υποθέσεων αφού έχουν εξατληφθεί τα εθνικά ένδικα μέσα. Εκτός αν εμείς πούμε ότι ε, οι εθνικές προσφυγές είναι αναποτελεσματικές. Αν το πούμε αυτό, τότε εμείς θα πρέπει να χειριστούμε αυτές τις 32.000 υποθέσεις. Και από τη δική μας πλευρά και από πολιτικής ε, σκοπιάς δεν είναι προφανές να πει κανείς ότι το συνταγματικό δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο ενός συμβαλωμένου κράτους, είναι αναποτελεσματικό και να το αποκλείσουμε ε, από όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Από νομικής πολιτικής πλευράς αυτό δεν θα ήταν δόκιμο. Έκτοτε βέβαια έχουμε ε, επιληφθεί στρατηγικών υποθέσεων και έχουμε δώσει αποφάσεις, παραδείγματος χάρη για την σύλληψη και κράτηση μέλους του ίδιου συνταγματικού δικαστηρίου. Αρπασλάν Ασλάν λέγεται αυτή η υπόθεση, αν η προφορά μου είναι σωστή. Επίσης, μια άλλη υπόθεση για την οποία αποφανθήκαμε, άρση ασυλίας, βουλευτικής ασυλίας ενός ε, μέλους του φιλικορδικού Κόμματος, ε, σύλληψη και κράτηση, το λόγο ε, βουλευτή, επομένως οι βουλευτοί δικαστές. Επίσης, είχαμε μια άλλη απόφαση που αφορούσε σύλληψη δημοσιογράφων μια άλλη που αφορούσε σύλληψη και κράτηση πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών και μια πέμπτη για ΜΚΟ. Άρα μέσα σε αυτές τις πέντε leading cases όπως τις λέμε, βασικές ε, υποθέσεις, είχαμε ε, τις πέντε βασικές ομάδες ε, θυγόμενων. Βουλευτές, δικαστές, ακαδημαϊκούς δημοσιογράφους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με βάση τις πέντε αυτές υποθέσεις προχωρούμε. Δεν σας κρύβω όμως πως πρόκειται για μείζωνα πρόκληση. Και, και γιατί την ανέφερα. Η χρήση του άρθρου 18 που προανέφερα. Ε, αφορά και την Τουρκία. Όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και την Τουρκία. Είναι λοιπόν πρόκληση βεβαίως και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας. Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη ε, χώρα ε, από την οποία έχουμε τόσα πολλά αιτήματα και προσφυγές 8.860 ε, κάτι υποθέσεις αφορούν την Τουρκία 15.000 αφορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία μετά είναι η Τουρκία, Ουκρανία, Ρουμανία κτλ με αυτή τη σειρά. σε ό,τι αφορά αυτό το living instrument, ζωντανό εργαλείο, το δόγμα αυτό και τις διαφορές ε, τις ε, κλιματικές. Πράγματι, χρειάστηκε να ασχοληθώ με το ζήτημα αυτό, διότι την προηγούμενη εβδομάδα με κάλεσαν ε, σε ένα πρόγραμμα εργασία, διότι η πρόεδρος Γεωργίας και πρόεδρο ε, τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, του Συμβουλίου τη Ευρώπη, έχουν βάλει προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή και τα κλιματικά ζητήματα. Πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το αδελφό αν θέλετε σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα το Συμβούλιο τη Ευρώπη να εργαστεί επί ε, της κατάρτισης ενός πληρωματικού πρωτοκόλου στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα αφορά ακριβώ το θέμα του περιβάλλοντο. Και θα υπάρξουν δύο μεγάλε διασκέψει για το περιβάλλον που οργανώνει η Γεωργιανή Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Η μία θα λάβει χώρα στι 27 Φεβρουαρίου και η δεύτερη στι 9 Απριλίου. Human Rights for the Planet, ανθρώπινα δικαιώματα για τον πλανήτη είναι ο τίτλο είναι ένας προκλητικός θα έλεγα τίτλος ε, που μένει στο μυαλό. Και είδα λίγο την ομολογία για να προετοιμαστώ, έφτιαξα και ένα θεματικό δελτίο όπως το λέμε για να δούμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την ομολογία και με έκπληξη διαπίστωσα ότι έχουμε περίπου 100 αποφάσεις ε, που άπτονται των ζητημάτων του περιβάλλοντος κατά το μάλλον ήτον, αφορούν την ιδιωτική ζωή, την προστασία ε, της ιδιωτικής σφαίρας όταν η ρήπανση αφορά την ε, ε, ιδιωτική ζωή και τη βιωσιμότητα. Λόπες Όστρα κατά Ισπανίας ήταν η πρώτη υπόθεση με την οποία ξεκίνησαν αυτές οι δικαστικές διαφορές και επίσης υπό το πρίσμα πολλών άλλων διατάξεων της Σύμβασης, δικαίωμα στη ζωή, η ελευθερία ενημέρωσης πληροφόρησης όταν υπάρχει ζήτημα ατμοσφαιρικής τύπας κτλ. κτλ. Πρόσφατα, το 2019, είχαμε και την υπόθεση Κορντέλα κατά Ιταλίας που αφορά ακριβώς ε, τις επιβλαβείς ε, ε, συνέπειες και πτώσεις της δουλειάς ενός εργαστήριου. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και θα ήθελα επίση να σας πω πως ε, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των κάτω χωρών που εμέσως αναφερθήκατε για το Δεκέμβριο του Ουτζέντα κατά... Λε, εκεί ήταν ε, πάλι μια σημαντική ε, υπόθεση για την ομολογία μας. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε αυτή την ομολογία χωρίς να έχουμε μια σύμβαση, σύμβαση στη δεσή μα που θα αφορά συγκεκριμένα το περιβάλλον. Γιατί άμεσα και το περιβάλλον δεν γίνεται λόγο σε καμία σύμβαση. Προσπαθήσαμε παρόλα αυτά και σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Να οικοδομήσουμε σιγά σιγά ένα ε, νομολογιακό κόρπους αρκετά ευρύ για τα θέματα του περιβάλλοντος. Φυσικά αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα πρόσθετο συμπληρωματικό πρωτόκολλο με διατάξεις ε, πολύ συγκεκριμένες, αυτό θα μας οδηγήσει στο να έχουμε μια πολύ πιο στέρεη βάση πάνω στην οποία θα αναπτύξουμε τη σχετική νομολογία. Για την κυρία Κάνκο. Θα σας ε, απογοητεύσω δυστυχώς από την έννοια ότι εκρεμεί αυτή τη στιγμή μια υπόθεση που αφορά το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε, αλλά δυστυχώς ε, ε επιφυλάσσομαι και δεν μπορώ να μιλήσω πιο εκτεταμένα για το θέμα αυτό, ε, λόγω εχεμήθειας. Και είναι μια σοβαρότατη υπόθεση. Θα τοποθετηθούμε ε, συντόμως. Σας ζητώ λοιπόν λίγη υπομονή. Και ε, δεσμεύομαι ότι το γραφείο μου θα σας ενημερώσει για την ετοιμιγορία. Γιατί άπτεται του ζητήματος ακριβώς ε, που θίξατε. για τους Ισπανούς κρατούμενους, Καταλανούς κρατούμενους το ισπανικό ζήτημα αυτό και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν ενδεχομένως ε, ε, για να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων. Ναι, πράγματι υπάρχει το άρθρο 34 της σύμβασής μας που ορίζει πως τα συμβαλόμενα κράτη υποχρεούνται να μην θέτουν εμπόδια, πόσο δε μάλλον πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα είναι προφανέ πω αν υπάρχει προσφυγή ε, που φτάνει ενώπιον του δικαστήριου και η οποία αναφέρει τέτοιου είδου προβλήματα, το δικαστήριο θα πρέπει να διαπιστώσει κατά πόσον ε, υπάρχει παράβαση του άρθρου 34. Και μάλιστα αυτό έγινε όταν ε, σε μια υπόθεση που αφορούσε ε, ένα σοφρονιστικό έδρυμα ε, να δούμε αν είχαν πρόσβαση, τη δυνατόν να έχουν πρόσβαση κρατούμενοι στο δικαστήριο. Το γνωρίζουμε δυστυχώς το πρόβλημα και το πλαίσιο αυτό και πράγματι έχουμε διαπιστώσει παράβαση του άρθρου αυτού κατά το παρελθόν. Θερμότατα για την ερώτησή σας. Περιμένουμε να βάλω τα ακουστικά. Ε, επιτρέψτε μου να μιλήσω στα ελληνικά, ε, μια και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ε, η ερώτησή σας είναι κέρια σημασίας αναβεσβήτητα και αφορά αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή την προσπάθεια εναρμόνισης των αρχών της σύμβασης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για το δικαστήριο. Στο δικό μου το τμήμα είναι και ο Βρετανός δικαστής. Ο Βρετανός δικαστής αποφαίνεται και γνωρίζει το common law, χρειάστηκε να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσω να καταλάβω τη δική του γλώσσα και εκείνος να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβει την δική μας νομική γλώσσα. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε κάθε μέρα να το επιτύχουμε. Είναι μια πρόκληση. Στο ίδιο τμήμα υπάρχει ο δικαστής από την Αρμενία και φέρνει όλες τις υποθέσεις της Αρμενίας. Υπάρχει ο δικαστής της Ανδόρας, ο οποίος φέρνει υποθέσεις που βασίζονται στο ρωμαϊκό δίκαιο, διότι πιστέψτε με, στην Ανδόρα του 21ου αιώνα για μεγάλα κομμάτια του δικαίου εφαρμόζεται το ρωμαϊκό δίκαιο και πάμε πίσω στους Ιουστινιάνιου κώδικες. Είναι απίστευτο αλλά αληθές. Πήγαμε σε επίσημη επίσκεψη στην Ανδόρα τον περασμένο Ιούνιο και το διαπιστώσαμε. Καταλαβαίνετε επομένως τι σημαίνει για ε, έναν ε, δικαστή να έχει μπροστά του όχι μόνο όλους τους κλάδους του εθνικού δικαίου αλλά και διάφορες νομικές ε, ένομες τάξεις. Ανέφερα το Ενώμανο Βασίλειο, την Αρμενία, την Ανδόρα, έχουμε τη Φιλανδία, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, την Τσεχία, την Πολωνία, στο ίδιο τμήμα πάντοτε Κανείς πρέπει να, μπορέσει να βρει μια κοινή γλώσσα με τους ε, συναδέλφους. Είναι κάτι το πραγματικά ε, δύσκολο στην καθημερινή ζωή του δικαστηρίου, αλλά το προσπαθούμε και είναι μια πραγματική ε, πρόκληση. Madame la Présidente, l'impact de la sortie des σε σχέση τώρα με την επίπτωση του Brexit, θα ήθελα να πω ότι για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιστεύω, ελπίζω, να μην υπάρχει αντίκτυπος. Ε, την προηγούμενη Πέμπτη δεχτήκαμε τις επίσκεψη ε, του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και των άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, των τεσσάρων δικαιοδοτικών οργάνων και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου μας είπε ότι δεσμεύεται ως προς την σύμβαση. Το Human Rights Act επιβάλλει στους Βρετανούς να λάβουν υπόψη όχι μόνο τη σύμβαση αλλά και την ομολογία του δικαστηρίου. Οι, οι Βρετανοί, και αυτό το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα, είχα προεδρεύσει στο σχετικό τμήμα, μπορούν λοιπόν να ερμηνεύσουν υπό την συσταλτική έννοια το περιεχόμενο της σύμβασης, αλλά και υπό την διασταλτική. Μπορούμε να μην συμφωνούμε πάντα μαζί τους, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται διάλογος μεταξύ δικαιοδοτικών οργάνων. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ε, δημιουργηθεί προβλήματα επί του παρόντος. Τώρα, ως προς την επίπτωση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση, θα ήθελα να πω ότι φυσικά θα είναι θετική για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, των νομοθεσιών. Δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως αποχρώσεις σε σχέση στο bis in idem για παράδειγμα, δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να δικαστεί δύο φορές για το ίδιο έγκλημα. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει μια κάπως διαφορετική ερμηνεία για το bis in idem. Πιστεύω ότι ε, έχει αποφανθεί και το, γνωρίζω ότι έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2010 επί του ζητήματος και νομίζω ότι η δική σας Επιτροπή θα μπορέσει στο μέλλον και στην περίπτωση προσχώρησης θα μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς την θέσπιση διαλόγου και με το δικό μας ε, δικαστήριο και με το δικαστήριο του Λουξεμβούρου. Εμεί είμαστε ανοιχτοί για ένα τέτοιο διάλογο. Σε σχέση με την πρόσβαση, με το δικαίωμα της άμβλωσης, είπαμε ότι ε, δυστυχώς δεν υπάρχει συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα μεθοδολογικά ε, δυστυχώς τα κράτη έχουν δικαίωμα εκτίμησης και ερμηνείας, ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης και ερμηνείας. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για την σύγκληση αυτού του περιθωρίου. Όταν λοιπόν καταλαβαίνετε δεν υπάρχει συνένεση και τα περιθώρια ερμηνείας και εκτίμησης είναι ευρύτατα. Το ίδιο ισχύει όταν διαπιστώσουμε ότι οι χώρες δεν μπορούν να συμφωνήσουν πανευρωπαϊκά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το περιθώριο ε, δεν έχει όρια. Το έχουμε πει και στην περίπτωση της Ιρλανδίας και σε άλλες υποθέσεις. Όταν υπάρχει κίνδυνος για την μητέρα ή για τη γυναίκα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση στην άμβλωση, δηλαδή να μπορεί να διακοπεί η εγκυμοσύνη και δικαστικά. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτό το καθολικό δικαίωμα. Υπάρχει και η σύμβαση Σεντάου σε σχέση ε, δηλαδή με τα δικαιώματα της γυναίκας που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θυμάμαι καλά, ε, ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών και από τα περισσότερα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί στο άρθρο 16 χρησιμοποίησαμε το άρθρο 16 ως έμπνευση όπου γίνεται ε, λόγος για το να μπορεί η γυναίκα να αποφασίσει για το χρονικό διάστημα μεταξύ μίας ή περισσότερων εγκυμοσυνών. Δηλαδή, θα πρέπει να κρίνει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για μία εγκυμοσύνη. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία, η οποία δεσμεύει τα κράτη-μέλη χρησιμοποιήσαμε αυτή την σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη και άλλα ε, ένδικα μέσα και λάβουμε υπόψη και τη σύμβαση των ε, Ηνωμένων Εθνών. Αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορώ να σας δώσω σε αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι ε, υπάρχει και κάποιο άλλο που θα ήθελε να, ε, να λάβει το λόγο. Ναι, εν συντομία. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν περιμένα να ακούσω σχόλιο για την τρέχουσα υπόθεση. Για γενικότερα σχόλια περιμένα να ακούσω για αυτό το θέμα που τίθεται ξανά και ξανά, γιατί πρέπει να βρούμε το σημείο ισορροπίας μεταξύ ε, της προστασίας ε, παιδιών από τη μία και την ασφάλεια των ατόμων εδώ ε, σε σχέση με γονεί που έχουν διαπράξει αδίκημα. Το σημείο ισορροπίας πρέπει να βρούμε μεταξύ της εθνικής κυριαρχίας, την ικανότητα και δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν τα ίδια για την ασφάλεια των πολιτών τους και ε, το θέμα αυτό το οικογενειακό. Δηλαδή, ε, εγώ γενικότερα θα ήθελα να τοποθετηθείτε για το ευρύτερο αυτό θέμα και όχι για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Η Πρόεδρος, Παραμένει το ερώτημα, είναι αυτό το οποίο εσείς ε, αναφέρατε για την, τον αντιτρομοκρατικό νόμο για τα ε, θύματα για αυτούς που έχουν υποστεί ε, τα επιπτώσεις από την κατάχρηση αυτού του νόμου είναι όντως η πρόκληση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα ασφαλείας. Το έχετε ήδη σχολιάσει κύριε Πρόεδρε, και κύριε Σιλιάνε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ θερμά για τις εξηγήσεις σας και για την πολύ εμπεριστατωμένη γνώση σας για τους διάφορους φακέλους, τις διάφορες υποθέσεις. Ήσταν πάρα πολύ καλά καταρτισμένος για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτη φορά έρχεστε στην Επιτροπή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε όμως και θα συνεχίσουμε μιλώντας για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωση στο σύνολό τη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ε, όλα αυτά βοηθούν στην εναρμόνιση των προτύπων και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε, και γενικότερα στο διεθνές στερέωμα. Μιλήσαμε πολύ για την πολυμερή προσέγγιση. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση της πολυμερούς προσέγγισης και θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα εξετάσουμε και σε αυτό το πλαίσιο της οικουμενικότητας και της πολυμερούς προσέγγισης. Απαντήσατε πάρα πολύ περιστατωμένα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τα μέλη που ήρθαν και μου έθεσαν ερωτήσεις. Η Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι η επόμενη συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας θα λάβει χώρα από τις 10 ως τις 6 στις 17 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες και στις 18 Φεβρουαρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 2.30 μέχρι τις 6.30. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και στο επανειδήν.